Οι χώρες ε, για τις οποίες πρόκειται στις συμφωνίες επανεισδοχής ε, τηρούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ποιε είναι οι συμφωνίε για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν υπογράψει. Πάντω πρέπει να υπάρχει ένα μηχανισμό παρακολούθηση για το πώ εφαρμόζονται αυτέ τι συμφωνίε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουμε τις συμφωνίες επανεισδοχής του ώστε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τελευταία παρατήρηση. Φαίνεται να υπάρχει έλλειψη διαφάνειας ε, όσον αφορά τη λειτουργία της πολιτικής επανεισδοχής. Κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται κυρίως στα διμερή πρωτόκολλα εφαρμογής που υπογράφουν και συμφωνούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ένωση με τρίτες χώρες. Μπορεί να μα εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η θέση αυτών των πρωτοκόλων. Είναι δημόσια έγγραφα, είναι έγγραφα τα οποία έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν ε, η Επιτροπή μας ζητήσει πρόσβαση σε αυτά τα πρωτόκολλα εφαρμογής. Θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίζουμε τι συμβαίνει μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει, παραδείγματο χάρη, φαίνεται ότι κάποιο κράτο μέλο, α πούμε η Σλοβακία, θα έχει 27 Απριλίου μία μυστική συνάντηση στο Κίεβο σχετικά με την υπογραφή μια συμφωνία επανεισδοχή για ένα πρωτόκολλο για ένα πρωτόκολλο εφαρμογής με την Ουκρανία. για μια χώρα όπως η Ουκρανία θα πρέπει να δείξει η Επιτροπή ιδιαίτερη προσοχή. Τι κάνει η Ουκρανία με τους ετούντες άσυλο. Λαμβάνει μέτρα εξαιρετικά σκληρά. Ευχαριστώ. Κυρία Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Μανσέρβη για την ε, παρουσίαση του μετά από αυτόν τον ε, αμφισβητούμενο απολογισμό της Κομισιόν. Να πω και εγώ μερικά χωρίς να είμαι επαναληπτική από αυτόν που είπαν οι συνάδελφοι και όπου χοντρικά συμφωνώ. Χαίρομαι που μετά από την εφαρμογή 12 συμφωνιών και 6 με διαπραγματευτική εντολή καταλήγουμε μετά από 7 χρόνια στην εφαρμογή μιας αξιολόγησης την οποία εμείς περιμένουμε εδώ και πολλά χρόνια. Καλή αργά παρά ποτέ όμως. Έχουμε λοιπόν εμείς αυτήν τη βάση που είναι σε ένα πλαίσιο που όλοι γνωρίζουμε εδώ αρκετά καλά, αλλά που αποτελεί και τον καμβά ως προς τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σχετικά με την Νότια Μεσόγειο έχω μία ερώτηση, μία ισορροπία που θύμισε η συνάδελφος ότι φαίνεται εδώ να είναι ένα κλείσμα με μουρουνέλαιο, όπως είπε η συνάδελφος. Έχουμε εδώ τις θεωρήσεις την πολιτική των θεωρήσεων, αλλά έχουμε μετά και τις μεγαλόστομες αρχές που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη ερώτηση που δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα, αλλά που καθένα καθένας φαντάζομαι την έχει κατά νου, είναι ότι κατά, την κατά τις συζητήσεις και μετά την ψηφοφορία, μετά από την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, επιμείναμε ιδιαίτερα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στην ανάγκη που υφίσταται να βασιστούμε στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και στις διεθνείς οργανώσεις όταν έχουμε μικτές οργανώσεις ε, επανεισδοχής για να μπορέσουμε να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και εγώ εδώ Παναλαμβάνω την ανάγκη του να συνεργαστούμε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ανεξάρτητες φυσικά, και, τις, ε, και να μπορέσουμε σε αυτό το πλαίσιο να, συμμετέχει, να συμμετέχουμε και το Κοινοβούλιο με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο κάθε φορά το Κοινοβούλιο να είναι παρόν σε αυτές τις μικτές επιτροπές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις όμως παρακολουθώντας από κοντά θα μπορούσαν για μένα και για άλλους συναδέλφους φαντάζομαι να αποτελέσουν τον φρουρό κατά των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ένα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και μετά η συνεργασία με τις τρίτες χώρες είναι κάτι το πολύπλοκο και μπερδεμένο και κάπου έχει ε, κουτσουρευτεί από αυτό το σύστημα η Κομισιόν έχει επαρκείς πληροφορίες και αξιόπιστα στοιχεία για να μπορέσει να κάνει αυτή την αξιολόγηση και να ελέγξει αυτό το οποίο κάνουμε. Ελέγχουν γιατί εδώ ε, ε, παίζεται η ζωή των ανθρώπων για τους οποίους ορίζεται το θέμα της επανεισδοχής. Και το θέμα κύριε Μανσερβίζη της ε, αναστολής, ε, της ε, προσωρινής αναστολής της συμφωνίας, διότι για να αναστείλουμε πρέπει να έχουμε επαρκή αξιόπιστα δεδομένα. Μία χώρα η οποία παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα το παραδεχτεί για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην προσωρινή αναστολή. Πώς μπορείτε εσείς να, περάσετε, να ξεπεράσετε αυτή την επιφανειακή εικόνα και να μπορέσετε να διαπιστώσετε την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να την αποτρέψετε. Ξέρουμε όλοι ότι είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Και τρίτο, για να είμαι γρήγορη και να μην μακρηγορώ, τι γίνεται με τις ε, διμερείς ε, συμφωνίες ας πούμε, τύπου Λιβύη, Ιταλία ή Ιταλία την Ισία στη Νότια Μεσόγειο. Έχουμε προχωρήσει σε αυτές τις συμφωνίες ε, επανεισδοχής με τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης. Ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαρητήρια για το μαύρισμα. Είναι καταπληκτικά τα Κανάρια νησιά. Βέβαια είναι μακριά από την Τινησία, από την Αίγυπτο και από τη Λιβύη. Οπότε θα παραμείνεις μαυρισμένος για πολύ καιρό. Διευθύντα, εγώ άκουσα, με άκουσα το... με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τοποθέτησή σου, λέει ο μιλητής. Εμείς συναντηθήκαμε στο παρελθόν για να συζητήσουμε για μια ειδική συμφωνία Ιταλίας-Λιβύης και εσύ τότε μου είχες πει, μου είχες δηλώσει ότι οι διμερείς συμφωνίες είναι σημαντικές λήψη κοινοτικών συμφωνιών οι οποίες βέβαια παραμένουν πολύ σημαντικές και ήμασταν μαζί και με άλλους ε, συναδέλφους ε, στην Λιβύη όπως ήσουν και εσύ ε, για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα κεφάλαιο στη Συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να έχουμε και κάτι και για τα εμπορικά κλπ. Αλλά τα πράγματα πήγαν όπως πήγανε. Τα κίνητρα είναι πολύ σημαντικά, η ρήτρα των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς υπογράψαμε τη νέα εντολή της Frontex πριν από μερικές εβδομάδες. Θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η βούληση της Κομισιόν σχετικά και όποιον ψηφίσαμε το Frontex εμείς διαπιστώσαμε ποιες ήταν οι αδυναμίες του παρά την ε, τεράστια δυνατότητα ε, σε, σε, ανθρώπινο δυναμικό, την ικανότητα του, βουλευ, του διευθυντή κτλ. 50 άτομα εργάζονται για την ε, Frontex, οι υπόλοιποι είναι αποσπασμένοι από τα κράτη-μέλη και μόνο το 1 τρίτο των κρατών μελών έχει δώσει την άδεια να συμμετέχουν. Εχθές έγινε το Συμβούλιο και φάνηκε ε, έντονα ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά, μια τεράστια απόσταση θέσεων στις 4 Απριλίου το Κοινοβούλιο εκφράστηκε μαζικά υπέρ της ε, Μάλτας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Κύπρου και στο Συμβούλιο είδαμε να βγαίνουν οι εθνικοί εγωισμοί. Εμείς ε, στην περίπτωση της Ιταλίας έχουμε τη συμφωνία με τη Λιβύη, με την Τινησία, αλλά εμεί τι μπορούμε να κάνουμε όμως όλοι μαζί. Διότι αλλιώς ε, θα γίνει ό,τι έγινε και στη Βεντιμίλια, όπου μετανάστες ε, γαλλόφωνοι εξάλλου θέλησαν να πάνε στη Γαλλία και δεν τους άφησαν. Εμείς δεν θέλουμε ανταγωνισμούς, δεν θέλουμε άχρηστες αντιπαραθέσεις, αλλά ζητώ σε σένα που έχεις εξουσία και είσαι σαφής αλλά φυσικά και στην Επίτροπο το ρωτάω αλλά τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη ούτω ώστε αυτή, το, αυτό το βαθμιαίο, το σταδιακό πρόγραμμα επαναπατρισμού να μπορέσει να ολοκληρωθεί από την Ιταλία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ε, τρία άτομα που θέλουν να πάρουν το λόγο και μετά θα έχουμε τις απαντήσεις του κυρίου Μανσαρβίση πριν έρθει η κυρία Σεσίλια Μάλστρομ για να μας μιλήσει για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου ΔΕΗ. Παρακαλώ λοιπόν ε, τα άτομα που θα λάβουν τώρα το λόγο να περιορίσουν τα σχόλιά τους ε, στις ερωτήσεις που θέλουν να θέσουν. Η κυρία Μπόσκορτ. Ευχαριστώ. Ναι, Σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα υπήρξαν πολλέ αντιρρήσει για το από το Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα με την αποστολή στο Πακιστάν, διότι ορισμένες διεθνές συμφωνίες ε, δεν υπογράφησαν. Εσείς στην εισαγωγή σας είπατε υπάρχει μια ρήτρα περιφρούρησης μετά στην πράξη πώς πραγματικά μπορούμε εμείς να προβλέψουμε ότι αυτές οι διατάξεις μπορούν να είναι σεβαστές. Δεύτερη ερώτηση για την Τουρκία. Παρά τις ε, διαπραγματεύσεις ε, που ολοκληρώθηκαν είπατε «Α, χρειάζονται περισσότερα κίνητρα» ούτως ώστε να είναι πιο αξιόπιστη διαπραγματευτική διαδικασία. Απ' την άλλη όμως Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολος ο διάλογος για τις βίζες. Δεν καταφέρατε τίποτα σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό δεν είναι εθαρρυντικό. Ε, Η κυρία Βερζά. Θα κάνω αυτό που θέλετε όντως κύριε Πρόεδρε Μόνο μερικές ερωτήσεις, γιατί όλα τα υπόλοιπα υπόθηκαν και θα είμαι ακριβής. Μιλάτε για ρήτρα αναστολή σε περίπτωση σε περίπτωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς το βλέπετε όμως εσείς όταν ξέρετε πάρα πολύ καλά για τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις άλλες συμφωνίες της Ένωση. Δείτε τις συμφωνίες μας με τη Λιβύη και με την Τινησία, εντελώς άχρηστα όλα αυτά και εσείς κάνετε έναν απολογισμό ο οποίος είναι αρκετά αρνητικός. Γιατί λοιπόν συνεχίζουμε να επαναδιαπραγματευόμαστε και μετά για τις αραβικές χώρες. Εγώ έρχομαι από μία χώρα που στις πολιτικές συνεργασίες που στις ε, συμφωνίες ε, σαν αυτή με ε, την Ισία Τι ρόλο παίζουν αυτού του είδους οι ρήτρε όταν έχουμε διαπραγματευτεί συμφωνίες με την κυβέρνηση Μπεναλή. μπορούμε να έχουμε μετά λέτε στοιχεία αξιόπιστα. Αυτές οι διαδικασίες είναι επιβλαβείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. και μετά αυτή αυτός ο όρος, αυτή η όροι που χρησιμοποιείται, κράτηση κτλ. Είναι κάτι που με εκπλήσει, θα ήθελα να ξέρω κάτι παραπάνω. Ο κύριος Μπρόγκς. Ευχαριστώ για τα άτομα που ε, επιστρέφονται με βάση την συμφωνία επανεισδοχής. Πρέπει να δούμε πώς, ποια θα είναι η μεταχείριση τις οποίες θα τύχουν. Τα άτομα αυτά πρέπει να μας ενημερώσουν, πρέπει να ξέρουν ε, ποια θα είναι η μεταχείριση της οποίας θα τύχουν. Θα πρέπει να υποβάλουν αποδείξεις. Και θέλω να ρωτήσω, έχουμε, έχει επιστραφεί κανείς με βάση τις συμφωνίες επανεισδοχής όταν είναι τόσο εύκολο να αποφευχθούν αυτές οι συμφωνίες και θα πρέπει ε, να υπόκεινται σε αυτές τις συμφωνίες επισδοχής μόνο εάν αποδεικνύουν ότι ε, ίσως δεν θα τύχουν κακής μεταχείρισης. Ο χρόνος μας είναι πολύ λίγος και τώρα ο κύριος Μανσερβίση θα προσπαθήσει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός των ερωτήσεων και θα σας παρακαλέσω λοιπόν να ε, μιλήσετε επί της ουσίας και να είστε πολύ συγκεκριμένος. Ευχαριστώ. Πρώτα ε, για τις ερωτήσεις που αφορούν τη σχέση ε, ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές ε, Συμφωνίες Προσδοχής και στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες. Εμείς στην έκθεσή μας παρατηρήσαμε ότι πολλά κράτη-μέλη προτιμούν τις διμερείς συμφωνίες από τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές συμφωνίες. Παρόλο που τα ίδια τα κράτη-μέλη είχαν ε, συζητήσει ε, με επιμονή αυτές τις ευρωπαϊκές συμφωνίες. Βλέπουμε Ε, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει μια απότομη μετάβαση από τις διμερείς ε, στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, απλά να μην συνεχίσουμε να, χρησιμοποιούμε μόνο τις διμερείς. Εάν θεωρείτε ότι εάν θεωρούν τα κράτη-μέλη ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιούν τις διμερείς συμφωνίες, τότε ας κάνουμε μία ε, ε, αξιολόγηση και να εξετάσουμε αυτά τα συμπεράσματα. Όταν δεν υπάρχουν ε, οι ευρωπαϊκές συμφωνίες, λέμε αυτό που είπαμε και, και πριν από μερικούς μήνες για τις ε, ε, συμφωνίες ανάμεσα στην Ιταλία και στη Λιβύη. Δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Συμφωνία, υπήρχε μια διμερή συμφωνία η οποία εφαρμοζόταν αποτελεσματικά. Όπως είχα πει και τότε, και η Ιταλία πάντα ακολουθούσε ε, αυτή την προσέγγιση, το καλύτερο θα ήταν να έχουμε μια ευρωπαϊκή συμφωνία και θα ήταν καλύτερο ε, η Ιταλία να κάνει τις διαπραγματεύσεις της με βάση μια ε, γενικότερη ευρύτερη ευρωπαϊκή συμφωνία. Όσον αφορά τις συμφωνίες, τις συμφωνίες που έχουμε τώρα με την Τινσία. εάν ε, μπορεί να αποδεχθούν και αυτές εξίσου αποτελεσματικές όπως και οι συμφωνίες με τη Λιβύη. Και η πρόκληση θα είναι να έχουμε μία ευρωπαϊκή ε, συμφωνία επενδυσδοχής με την Τινησία. και θα χρησιμοποιήσουμε την, τις εμπειρίες ε, με βάση ε, τα, το, τα συμπεράσματα που θα έχουμε στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, Εσωτερικών Υποθέσεων κτλ. Θα συζητήσουμε ποια είναι η δυνατότητα για να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια συμφωνία επανεισδοχής με την Τινησία. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε οι ε, επιστροφές που γίνονται με βάση, ε, διμερείς, με βάση τις διμερείς συμφωνίες να είναι αποτελεσματικές. Μπορεί ο Frontex να παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο. Θα έλεγα ότι η εκτέλεση των ε, συμφωνιών επανεισδοχής είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Μπορούμε όμως να συζητήσουμε έναν πιο ενεργό ρόλο του Frontex όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών. Όσον αφορά τώρα την, την τεκμηρίωση, σε κάθε συμφωνία υπάρχει ένα άρθρο που προβλέπει ότι αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα από την χώρα καταγωγής, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκδώσει ένα ταξιδιωτικό έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει την επιστροφή του ατόμου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, βοηθάει στην έκδοση αυτών των εγγράφων. Για το ερώτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρθηκε πολλές φορές από την εφαρμογή ε, των συμφωνιών μάθαμε ότι πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να έχουμε ένα καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε πολλές πληροφορίες από την κοινωνία των πολιτών, από τις ε, διεθνείς οργανώσεις, από ε, τις δικές μας εκπροσωπείες στις χώρες και βασιζόμαστε σε όλη αυτή την πληροφόρηση. Πρέπει όμως να έχουμε έναν μηχανισμό παρακολούθησης, να έχουμε μία ρήτρα αναστολής και να έχουμε και κίνητρα ε, για τη δημιουργία αυτού του συστήματος, όπως αυτό που κάνουμε τώρα στο Πακιστάν. Και επιπλέον πρέπει να συνοδεύσουμε τις επιστροφές με μέτρα που θα επιτρέπουν τις χώρες υποδοχής να ε, εντάξουν καλύτερα τα άτομα που επιστρέφουν. ω τώρα ήταν σαφέ ότι ε, χρησιμοποιούσαν την επανεισδοχή ω αντιστάθμισμα, για τι ε, συμφωνίε διευκόλυνση θεωρήσεων και εφόσον έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι συμφωνίες διευκόλυνσης θεωρήσεων, πρέπει να ε, ενισχύσουμε και τις συμφωνίες επανεισδοχής λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να έχουμε όμως και ενημέρωση και κατάρτιση των συναριοφυλάκων. Και φυσικά θα συνεχίσουμε αυτή την κατάρτιση. για τα διμερεί πρωτόκολλα τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε, κυρία Ουατάλα, τίποτα για κανένα κρυφό ε, ε, μυστικό πρωτόκολλο. Δεύτερον, για τα πρωτοκόλλα που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και υπάρχουν και στις μικτές, επιτροπής, ε, επιτροπές μπορείτε να απευθυνθείτε στα κράτη-μέλη αλλά και σε εμάς και μπορούμε λοιπόν να σας παρέχουμε αυτά τα έγγραφα. Τα περισσότερα πρωτόκολλα από όσο γνωρίζουμε αφορούν κάποιες λεπτομέρειες για το σημείο εισόδου Εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα για μυστικά τμήματα ή μυστικά περτόκολλα. Για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Είναι και αυτό μία από τις συστάσεις μας στις μικτές ε, επιτροπές θα θέλαμε να ανοίξουμε τη συμμετοχή στις ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στις διεθνείς οργανώσεις έτσι ώστε να λάβουμε ε, τη δική τους γνώση και να προετοιμάσουμε την εφαρμογή αυτών των ε, συμφωνιών. Η Επίτροπος ε, Μάλστρομ είναι ήδη εδώ. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να κλείσω συνοπτικά λέγοντας ότι αυτή είναι μια πρώτη έκθεση ε, ε, η οποία έγινε εφόσον ζητήθηκε από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης αλλά χρειάζεται χρόνος για να το αξιολογήσουμε αυτό, να δούμε το πλαίσιο Και το, το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε μόνο συμφωνίες επανεισδοχής. Μπορούμε να έχουμε ίσως μια εταιρική σχέση κινητικότητας. Κάτι που θα αποτελούσε ένα μέρος των προϋποθέσεων. Πρέπει επίσης να δούμε και ε, ευρύτερα όλη την ε, πολιτική προσέγγιση, την πολιτική για τις επιστροφές. Έχουμε μια νέα οδηγία ε, περί επιστροφών που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή και πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί ως τώρα η ευρύτερη πολιτική ε, επιστροφών, της οποίας ε, οι συμφωνίες επιστροφής είναι μόνο ένα ε, στοιχείο. Η κυρία Μάλστρομ μπορεί σίγουρα να απαντήσει πολύ καλύτερα σε όλα σας τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις εντατικές προσπάθειες που κάνατε να συνοψίσετε την αξιολόγηση για τις συμφωνίες επανεισδοχής. Σας ευχαριστούμε και ετοιμαζόμαστε λοιπόν να προχωρήσουμε και να υποδεχθούμε την ε, Επίτροπο κυρία Σεσίλια Μάλστρομ και να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημέρης της διάταξης. Ναι, ναι,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 Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την Επίτροπο Μάλτσον που ήρθε στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα από το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων. Και ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι η συνεδρίαση που κάναμε μόλις προηγουμένως και κλεισμένων ε, των θυρών ξεκίνησε με το ότι εκφράσαμε τη λύπη μας ε, για την ε, τρομοκρατική επίθεση που έγινε χτες στο Μίσχ στη Λευκορωσία. Εκφράζουμε λοιπόν την θλίψη μας για τα θύματα και Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επαναλάβουμε τώρα που βρισκόμαστε στην όλο μελή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ξεκινάμε δίνοντας το λόγο στην Επίτροπο Σεσίλια Μάλστρομ για να μας μιλήσει για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΔΕΗ. Κύριε Μάλστρομ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι και πάλι κοντά σας. Σχεδόν κατευθείαν έρχομαι από το Λουξεμβούργο μετά από μια συνεδρίαση δύο ημερών του Συμβουλίου δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων. Θα σα πω λοιπόν ποιε είναι οι τελευταίες εξελίξεις, θα σας πω ποια είναι τα θέματα στην μέση διάταξη τη Επιτροπής και θα είμαι διαθέσιμη και για τι δικέ σα ερωτήσει και σχόλια. Όπω φαντάζεστε, η κύρια συζήτηση χθε αφορούσε τα θέματα της μετανάστευσης στην Νότια Μεσόγειο. Έγινε μια μακρά συζήτηση από το θέματος αυτού χθε. Όπως φαντάζομαι ότι θα γνωρίζετε, γιατί έστειλα μια επιστολή προς τον πρόεδρό σας, έστειλα ε, μια επιστολή προ τον επικεφαλή του Συμβουλίου των Υπουργών, εξηγώντα τι ακριβώ κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τη ροή μεταναστών, ε, τι κάνουμε όσον αφορά τι δραστηριότητε ε, του οργανισμού Frontex, πώ βοηθάμε του ανθρώπου επιτόπου Παρουσίαζε επίσης ε, και τις ανάγκες για πρόσθετη χρηματοδότηση και ζητούσε αλληλεγγύη από τα κράτη-μέλη για τους ανθρώπους αυτούς ε, που βρίσκονται αποκλεισμένοι στην Τινησία, στην Λιβύη, στα σύνορα με την Αίγυπτο, καθώς και για τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη. Η επιστολή περιλαμβάνει επίσης και ε, μια σύντομη σύνοψη των ταξιδιών μου στην την Ισία και στην Αίγυπτο ε, και σχετικά με τις προσπάθειες ε, για ένα διάλογο για τα θέματα κινητικότητας ε, με τις χώρες αυτές. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο πολλοί από εσά θα ήσασταν παρόντες στην συζήτηση και θα αναγνωρίζετε τα στοιχεία της συζήτησης τα οποία και εκεί συζητήθηκαν. Τονίσαμε την ανάγκη για αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάγκη να ενισχύσουμε τον οργανισμό Frontex και χαίρομαι διότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, δηλαδή όχι μόνο να έχουμε μια ενότητα ε, των συμπεράσματων του Συμβουλίου, αλλά να έχουμε μια παράταση του πιλωτικού προγράμματος της Μάλτας. Και αυτό έγινε αποδεκτό. Όπως ξέρετε, η Μάλτα πλήγεται ιδιαίτερα, πλήττεται ιδιαίτερα από ε, αυτές τις κινήσεις τις μεταναστευτικές. Ε, η Μάλτα είναι μια πολύ μικρή χώρα και έφτασαν πάνω από άτομα ε, στις ακτές της Μάλτας. Η Μάλτα έχει πολύ περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης και χαιρόμαστε που παρατείνεται αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Πολύ λίγα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν ότι δέχονται να πάρουν ε, μετανάστες από τη Μάλτα. Η Γερμανία δέχτηκε να πάρει 100 άτομα. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι έχουμε παράταση του προγράμματος. Επίσης, συζητήσαμε και την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του οργανισμού Frontex. Ελπίζουμε ότι μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, καταλήξουμε σε μεταρρύθμιση του κανονισμού Frontex. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουν ε, οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επόμενη συνεδρίαση στις 12 Μαΐου θα συζητήσουμε και πάλι αυτά τα θέματα και πάλι στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκεται η κατάσταση στην Νότια Μεσόγειο και ελπίζω θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και τα γενικότερα θέματα πολιτικής μετανάστευσης. Στα τέλη Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσουμε το θέμα της μετανάστευσης για να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση του Συμφώνου Μετανάστευσης που ξεκίνησε επί Γαλλικής Προεδρίας και θα γίνει μια γενική συζήτηση για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά την μετανάστευση και την ένταξη. Θα επανέλθω όμως σε αυτό το θέμα λίγο αργότερα. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι από τα χθεσινά μας συμπεράσματα. Σαφώ υπάρχει ανάγκη αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν και η συνάδελφος κυρία Τζορτζίεβα παρούσα για να εξηγήσει ε, πώ ε, βοηθούν οι δικέ της μονάδε και στην Τινησία και στην Αίγυπτο και μα έδωσε μια πλήρεστερη εικόνα του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην Νότια Μεσόγειο. Επίσης, ε, μετά το γεύμα έγινε και μια δύσκολη συζήτηση για το θέμα των καταλόγων ονομάτων επιβατών ε, του PNR. Πρότεινε ε, ε, κάτι το Φεβρουάριο Επιτροπή όπου υπάρχουν σημαντικές τροποποίησεις μετά τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή η πρόταση αυτή είναι διαφορετική από την πρόταση του 2007. Είναι πιο περιορισμένο το πεδίο εφαρμογή ε, και το γεωγραφικό πεδίο. Μιλά μόνο για τι πτήσει ε, από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλά για την προστασία των δεδομένων και συμπεριλαμβάνει και ένα άλλο στοιχείο καινοτομία ότι τα δεδομένα θα πρέπει να φυλάσσονται σε μία ανώνυμη βάση δεδομένων μετά την πάροδο ενός μηνός και μόνο ε, κατά περίπτωση μπορούν να εξετάζονται οι διάφορες υποθέσεις. Έγινε μία μακρά συζήτηση, είχε γίνει ούτως ή άλλως συζήτηση στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και πολλές χώρες, η πλειοψηφία των χωρών, επιθυμούν να συμπεριλαμβάνεται και ένα ενδοευρωπαϊκό PNR. Η Προεδρία είχε εξετάσει διαφορετικέ εναλλακτικέ λύσει για το χειρισμό αυτού του θέματο. Μία εναλλακτική λύση είναι το να μην συμπεριλαμβάνονται οι ενδοευρωπαϊκέ πτήσει δεύτερη εναλλακτική λύση ήταν προαιρετική συμπερίληψη κάποιων ενδοευρωπαϊκών πτήσεων σε συγκεκριμένα δρομολόγια. Τρίτον, υποχρεωτική συμπερίληψη κάποιων ενδοευρωπαϊκών πτήσεων. Και τέταρτον, υποχρεωτική συμπερίληψη όλων των ενδοευρωπαϊκών πτήσεων. Έγινε μια, ένας γύρος και τα περισσότερα κράτη-μέλη προτίμησαν τη δεύτερη εναλλακτική λύση, δηλαδή προαιρετική συμπερίληψη ορισμένων ενδοευρωπαϊκών πτήσεων. Κάποια κράτη-μέλη εξέφρασαν υποστήριξη τουλάχιστον μακροπρόθεσμα να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά όλε οι ενδοκινοτικέ πτήσει και κάποια, μειοψηφία υποστήριξε και την πρόταση τη Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει ε, το να συλλέγονται δεδομένα PNR για όλες τις πτήσεις, ε, αλλά ε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει αυτή τη στιγμή και επομένως προτείνουμε μια σταδιακή προσέγγιση για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το μέτρο τελικά και να αποκτήσουμε την εμπειρία συλλογής δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν και στοιχεία κόστους που δεν πρέπει να παραμελούμε και σε σύγκριση με τι Ηνωμένε Πολιτείε, πρέπει να δούμε ότι και εκείνοι ξεκίνησαν με τι εξωτερικέ πτήσει πρώτα πριν περάσουν στην καταγραφή δεδομένων και για τι ε, πτήσει εντό των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συνεχιστεί η συζήτηση του θέματο και θα είναι πολύ χρήσιμο για μα να ακούσουμε τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζω ότι δεν θα είχατε προφανώ ε, ακόμη την ευκαιρία να συζητήσετε αυτό το θέμα αλλά αν έχετε σχόλια μπορείτε και τώρα να μου υποβάλλετε τις πρώτες σας παρατηρήσεις. Όπως πάντοτε στην ημερήσια διάταξη υπήρχαν τα θέματα του CIS και του VIS και στρέφω το βλέμμα προς τον κύριο Κοέλιο γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Όλα προχωρούν σύμφωνα με το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή το VIS σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τον Οκτώβριο του 2011 περιμένουμε κάποια πρόοδο σε σχέση και με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ε, και για το ΣΥΣ 2 ε, επίσης υπάρχει η αναμενόμενη πρόοδος. Υπάρχουν δύο κίνδυνοι εδώ. Υπάρχει ένα θέμα του αν θα είναι ε, τα κράτη-μέλη έτοιμα και το δεύτερο ερώτημα αφορά την ετοιμότητα από το, να περάσουμε από το CIS 1 στο CIS 2. Ε, Αυτού του κινδύνου ε, σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών θα προσπαθήσουμε να του μετριάσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν. Ε, συνεχίζουμε επίσης τις διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε κάποια πιο οριστικά αποτελέσματα με τον τριμερή διάλογο. Ε, γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ Εστονίας και Γαλλίας. Έγινε επίσης μια συζήτηση για τη διαδικασία του ΠΡΟΥΜ, ε, κατά τη διαδικασία του μεσημεριανού γεύματος. Στις 26 Αυγούστου νομίζω ότι έχει τεθεί η προθεσμία και τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσουν να τηρήσουν αυτή την προθεσμία. Πάντως ε, ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού βρίσκονται τα κράτη-μέλη και κάποια κράτη-μέλη πρόσφεραν τεχνική βοήθεια και υποστήριξη προς άλλα κράτη-μέλη. Ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια κονδύλια και για προκηρύξεις για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να είναι ε, σε επιχειρησιακή ετοιμότητα κάτι που θα μας βοηθήσει για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Συζητήθηκε επίσης ε, και το θέμα του προγράμματος δράσης ε, της Ελλάδας που έχει προχωρήσει και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε σε ε, όλα τα Συμβουλία Υπουργών ΔΕΗ. Στο πλαίσιο των, της συνεδρίας των Υπουργών Δικαιοσύνης, σήμερα το πρωί παρακολούθησε τα πρώτα δύο σημεία. Η Επίτροπος Ρέντινγκ φαντάζομαι θα σας ενημερώσει για τα υπόλοιπα σημεία. Το πρώτο θέμα ήταν μια σύντομη ενημέρωση για την οδηγία για την ε, σεξουαλική βία κατά των παιδιών. Έγινε μια συζήτηση για τις ε, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφορικής. Δεν ήταν εύκολη η συζήτηση στο Συμβουλίο γιατί διαφέρουν οι απόψεις των κρατών μελών όσον αφορά τα διαθέσιμα μέσα. Η Προεδρία προσπαθεί να καταλήξει σε συμβαστικές λύσεις. Γίνονται ακόμη συζητήσεις για το επίπεδο των κυρώσεων, για τις επιβαρυντικές συνθήκες και για τα σημεία στα οποία ε, υπάρχουν δυσκολίες. Πριν από δύο εβδομάδες έγινε επίθεση και κατά ε, της Επιτροπής ε, στο διαδίκτυο και στο Κοινοβούλιο και είμαστε σε γρήγορση όσον αφορά τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και ετοιμάζουμε τα κατάλληλα μέτρα. Η οδηγία του 2005 δεν είναι μια επίκαιρη οδηγία και σαφώς ε, χρειάζεται ένα μήνυμα ότι είναι επίγοντα αυτά τα θέματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και αύριο η Ουγγρική Προεδρία οργανώνει στην Βουδαπέστη ένα σχετικό συνέδριο. ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια ε, συμφωνία επί του θέματος πριν το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να αναφέρω και κάποια σημεία ακόμη για να σας παρουσιάσω το σύνολο των θεμάτων. Ένα θέμα που συζητήθηκε εν συντομία χθε και συζητήθηκε και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο είναι το θέμα του κοινού συστήματος ασύλου. Στο Συμβούλιο συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση και θα ήθελα να σας ενημερώσω επί του θέματο. Η δημιουργία μιας κοινή πολιτικής ασύλου ίσως είναι τώρα περισσότερο επίγουσα παρά ποτέ. το να έχουμε όλες τις συμφωνίες μέχρι το 2012 νομίζω ότι είναι εφικτό και πιστεύω ε, και είμαι ευτυχής διότι η Πολωνική Προεδρία συμμερίζεται την άποψη αυτή και θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να το καταφέρουμε. Πρέπει να διαμορφώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία για την προστασία στην Ευρώπη. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για τους ετούντες άσυλο που φτάνουν στην Ευρώπη αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εθνικές μας διοικήσεις. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων από τα κράτη-μέλη με αποτελεσματικό τρόπο γιατί όλο και περισσότερο έχουμε μικτές ροέ, όπως βλέπετε από, τις, από, τα, από τα πρόσφατα γεγονότα. Πρόσφατα είχαμε αρκετές εξελίξεις, ε, η οδηγία για τους κατοίκους ε, μακράς διάρκειας που επισήμως χθες ε, εγκρίθηκε, ψήφισε το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα με βάση την έκθεση Κιγιόν και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει ε, για την οδηγία για τα προσόντα. Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της Άνοιξης προσπάθησε μαζί με τα κράτη-μέλη να δει πού βρίσκονται οι δυσκολίες, πού βρίσκονται τα βασικά προβλήματα και σε συζήτηση με τους συζητητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προτείνουμε τροπολογίες και στην οδηγία για ε, την υποδοχή και στην οδηγία για τις διαδικασίες. Αυτό ελπίζω ότι θα βοηθήσει τις ε, συζητήσεις και θα υποβάλουμε αυτές τα στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο για να έχουμε μια συνολική συζήτηση για το πακέτο του ασύλου αρχές Ιουνίου θα το συζητήσει και το Σώμα των Επιτρόπων. Κάτι ακόμη και πιο σημαντικό είναι ότι θα διαμορφώσουμε μία ανακοίνωση για την ενδοκινοτική αλληλεγγύη. Η συζητήθηκε χθε και μέσα στο 2011 θα συζητηθεί εις βάθος. Κάτι το οποίο τόνισα και προς το Συμβούλιο χθε είναι ότι καλό όλους να προσπαθήσουν να αναζητήσουν μία λύση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγκατάστασης και θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα θεσμικά όργανα που έχουμε στη διάθεσή μας. Σίγουρα χρειαζόμαστε το πρόγραμμα επανεγκατάστασης ε, επιγόντως. Για την μετανάστευση έχουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020. Είναι σημαντικό για την μετανάστευση αλλά και για την εικόνα που θέλουμε να δώσουμε ε, στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε ένα οχυρό στο οποίο δεν δεχόμαστε νόμιμη ε, μετανάστευση. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό από οικονομικής, η πολιτικής ε, και κοινωνικής άποψης και πρέπει να έχουμε κάποια βασικά κριτήρια. Αυτή είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Στην Ολομέλεια του Μαρτίου είδαμε ότι είχαμε διαφορές ανάμεσα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά ελπίζω ότι θα εργαστούμε για να βρούμε λύση σε αυτές τις διαφορές. Επίσης, ελπίζω ότι θα έχουμε ε, πρόοδο τους ε, για την οδηγία των, για τις μεταθέσεις που γίνονται επιχειρησιακώς. Επίσης, Θέλουμε να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική και να δώσουμε ευκαιρία ε, στους νόμιμους μετανάστες. Γι' αυτό θα παρουσιάσουμε στις αρχές του Μαΐου μία ανακοίνωση για τη μετανάστευση και στις 24 Μαΐου θα έχουμε μια ετήσια έκθεση για το ε, άσυλο και τη μετανάστευση και την μετανάστευση των υπηκών τρίτων χωρών. Αυτές οι προτάσεις θα παρουσιαστούν και σε εσά και είναι πολύ ε, σημαντικές προτάσεις για τη συζήτηση ε, που θα γίνει τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη μετανάστευση. Αυτές οι προσπάθειες θα ολοκληρωθούν στο τέλος του χρόνου, μάλλον τον Νοέμβριο, με μια γενική προσέγγιση για τη μετανάστευση. Αυτό θα είναι ένα μήνυμα για τη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οποία θέλει να έχει μια συνεκτική και ισορροπημένη προσέγγιση για τη μετανάστευση. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν νέοι εσωτερικοί και εξωτερικοί στόχοι. Ανυπομονώ να ακούσω και τις δικές σας απόψεις και φυσικά είναι σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο να δούμε και τις εταιρικέ σχέσεις κινητικότητας που θα αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με την, την και την Αίγυπτο. Τέλος, για την εσωτερική ασφάλεια, όπως γνωρίζετε, με βάση τα συμπεράσματα καλωσορίζουμε την ε, στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μία πρώτη ετήσια έκθεση για τις δράσεις που έχουν αναλυφθεί. Θα είναι κοινή ε, ατζέντα, ε, επομένως ανυπομονώ και θα καλωσορίσουμε όλες τις δικές σας απόψεις. Θα έχουμε και ε, δύο ακόμα εκθέσεις για το οργανωμένο έγκλημα και την καταπολέμηση του, της τρομοκρατίας για το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να δούμε και τις ε, πτυχές που αφορούν την οικονομία. Πρέπει να προστατεύσουμε την νομική, ε, την νόμιμη οικονομία και θα, πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό για την παρακολούθηση της διαφθοράς και τις κατασχέσεις, έτσι ώστε το εφιστάμενο πλαίσιο να γίνει πιο ε, ισχυρό. Θα προτείνουμε ένα πακέτο τον Ιούνιο και το φθινόπωρο θα ε, έχουμε την πρόταση για τις κατασχέσεις. Ο στόχος είναι να έχουμε τις καλύτερες πρακτικές και να ενθαρρύνουμε την ε, μάθηση από μοτίμους και θα ε, πρέπει να σημειώσω ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ οι δηλώσει που είχαμε από το, Συμβούλιο Υπουργών του προηγούμενου Μαΐου. Τέλος, την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, ε, υιοθετήσει μια ανακοίνωση για την οδηγία για την κράτηση των προσωπικών δεδομένων. Εδώ θα συμπεριλάβουμε και ανησυχίε που είχαν εκφραστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ξεκινήσουμε μετά ε, συζητήσεις, θα έχουμε μια τεχνική ενημέρωση για εσά την επόμενη εβδομάδα και φυσικά μετά την έγκριση της ανακοίνωσης θα σας τη στείλουμε άμεσα. για τα ΕΦΗ e σύνορα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, ξεκινήσουμε ε, συζητήσεις και να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των ε, τεχνολογικών πρόοδων που έχουμε επιτεύξει. Αυτά λοιπόν για, από το Συμβούλιο και κάποια από τα στοιχεία που θα ακολουθήσουν Ανυπομονώ λοιπόν να συνεργαστώ και μαζί σας και περιμένω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ την κυρία Πίτροπο για την παρουσίασή της. Ήταν ιδιαίτερα λεπτομερής, ε, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο που είχαμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχω εδώ ένα κατάλογο με 14 ε, μέλη που θέλουν το λόγο. Σας λέω λοιπόν εξ αρχής να μην ε, ζητήσουμε περαιτέρω ε, ανοχή από τους διερμηνείς και γι' αυτό να περιοριστείτε στα σχόλια κατά τον τρόπο ε, που ε, έκανε και η κυρία Μάλστρομ και να αναφερθείτε στα θέματα που, τα οποία έθιξε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ε, για την κατάσταση στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα για τη μετανάστευση. Κυρία Επίτροπε, ξέρετε ότι θαυμάζω την προσωπική σας δέσμευση. Όμως ε, δεν είμαι ικανοποιημένο με το επίπεδο αλληλεγγύη που έχουμε έω τώρα. Δεν θα μιλήσω για αλληλεγγύη, αλλά για την έλλειψη αλληλεγγύη και για τι επιπτώσει αυτή τη έλλειψη. Έχουμε εντάσει ανάμεσα σε μεμονωμένε χώρε, ανάμεσα στου πληθυσμού, ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα επίσης συχνά έχουμε δηλώσεις ε, που συνδέονται με ακροδεξιά κόμματα. Αυτό δημιουργεί ε, πρόβλημα για τα ε, κόμματα που βρίσκονται στο μέσο και επίσης δημιουργεί πρόβλημα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε ένα πλοίο 47 ε, ναυτικά μίλια από τη Μάλτα και 45 από την Λαμπαντούσα. Τελικά δηλαδή ήταν δύο, κατά δύο μίλια πιο κοντά στη Μάλτα. Εδώ δημιουργούμε δηλαδή μη απαραίτητες εντάσει και θα θέλαμε αυτό να αλλάξει. Επίσης θέτουμε σε κίνδυνο ζωέ. Ξέρετε ότι ε, χάθηκαν 200 ζωέ την προηγούμενη εβδομάδα και έκτοτε τίποτα δεν έγινε πιστεύω ότι όλοι φέρουμε ε, τη ευθύνη για αυτές τις ζωές που χάθηκαν. Και τέλος, υπάρχει έλλειψη της, της Ευρώπης της προβολής της Ευρώπης. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι τραγικό και απορρέει από την έλλειψη της αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρετε ότι ε, έχει ενθαρρύνει την οδηγία 55 του 2001. Υπάρχει έλλειψη ε, υποστήριξη στο Συμβουλίο, αλλά θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μεγαλύτερη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την αλληλεγγύη. Ανησυχώ όμως εάν για την επέκταση ενός συστήματος που το οποίο εφαρμόζει εθελοντικά μία χώρα ε, σε άλλες χώρες. Ίσως αυτό να μην λειτουργήσει. Κάποιες, κάποια χώρα είπε ότι ε, θα πάρει 12 άτομα από τη Μάλτα. κάποια άλλη χώρα είπε ότι θα πάρει μια οικογένεια. Έχω αμφιβολίες για το αν θα μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Λόγω της προαιρετικής φύσης αυτού του προγράμματος εξορισμούς, εξορισμού ένα προαιρετικό πρόγραμμα σημαίνει ότι δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη σημαίνει ότι μια άλλη χώρα έχει την ευθύνη και απλά μια άλλη χώρα προτείνει εθελοντικά να την βοηθήσει. Υποστηρίζω βέβαια την ε, ε, τη δήλωση που μόλις κάνατε για μια επερχόμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τέλος, Είμαι περήφανος για τη χώρα μου που ε, προσπαθεί να σώσει άτομα ε, που κινδυνεύουν από πνιγμό. Όμως για μένα το να είμαστε Ευρωπαίοι σημαίνει να είμαστε και αλληλεγγύοι και ως τώρα είναι κάτι που δεν έχουμε δείξει. Ευχαριστώ κύριε Μπουσούτιλ. Μιλήσατε επί της ουσίας και μιλήσατε ξεκάθαρα και ελπίζω ότι και τα υπόλοιπα μέλη θα ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα. Η κυρία Γκέντς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τις πληροφορίες που μας δώσατε και έχω ορισμένα σχόλια και ερωτήσεις ε, για την κατάσταση στη Νότια Μεσόγειο. Γιατί αυτό είναι το ε, ε, κύριο θέμα, αν και μας μιλήσατε και για πολλά άλλα θέματα, εξίσου σημαντικά αλλά όχι τόσο επίγοντα. Υποστηρίζω και εγώ αυτά που μόλις είπε ο Σάιμον, διαβάζοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου δεν δόθηκε ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης. Μιλά για μια εθελοντική βάση και εδώ ε, τίθεται θέμα προθυμίας των χωρών να συμμετάσχουν στην παράταση του πιλωτικού προγράμματος. Ακόμη ε, συζητήθηκαν και κάποια πρόσθετα κονδύλια, κάποιοι πρόσθετοι πόροι. Έχει φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξουν κάποια κονδύλια, είναι πρόθυμα τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι επαρκής η πόρη αυτή τη στιγμή. Και πάλι διαβάζοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, βλέπω πολλά για τον έλεγχο των συνόρων, για τη συνεργασία σχετικά με την επανεισδοχή, σχετικά με τις κοινέ περιπολίες με την, την Ισία και πολύ λιγότερα για πραγματικούς πρόσφυγες από τη Λιβύη. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση. και η Μάλτα και η Λαμπεντούζα επίσης είναι ένα επίγον θέμα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν όχι μόνο το θέμα του ελέγχου αλλά και το θέμα των προσφύγων, το θέμα του ασύλου. Ακόμη είπατε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει μια πρόταση για τους οργανισμούς επιβολής ε, της νομοθεσίας και ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο διαφωνούσε. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη συμφωνία αυτή γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που θα αμφισβητηθεί και ενδεχομένως θα αντιτεθούμε σε αυτό. Ακόμη ε, για τις τροπολογίες που αφορούν τη μεταρρύθμιση του οργανισμού Frontex. Θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο. Αυτά προς τα παρόν γιατί ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Γκάντση, κυρία Δίκστρο. Εγώ φυσικά στη Σουηδία Επίτροπο, θα μιλήσω σου ειδικά. Σα ευχαριστώ για τη σαφήνειά σου, για το γεγονό ότι παρουσίασε τη στρατηγική, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα για τη μετανάστευση κλπ. Που μας ανέφερες και τα τελευταία δραματικά γεγονότα στη Βόρεια Αφρική. Όλα αυτά είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν συλλογικά και αλληλέγγυα από όλα τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται αλληλεγγύη και στα νότια σύνορα της Ευρώπης. Αλληλεγγύη που δοκιμάζεται μέρα με τη μέρα. Εδώ και μερικές εβδομάδες συζητιέται για το πώς θα ενεργοποιηθεί αυτή η οδηγία Και συζητάμε συνεχώς και ξανασυζητάμε, αλλά σε τι πλαίσιο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εχθές ε, έγινε μία ανακοίνωση και εσείς είπατε «Α, είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξεκινήσει αυτός ο μηχανισμός». Ε, Αλλά αυτή η οδηγία ξεκίνησε στην εποχή του πολέμου της Ιουγκοσλαβίας όπου είχαμε χιλιάδες άτομα που είχαν ε, επίγους ανάγκη προστασίας. Και σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πολλά κράτη-μέλη, δικά μας κράτη-μέλη δοκιμάζονται. Η Γερμανία υποδέχτηκε καμιά κατοσταριά άτομα αλλά ποιες άλλες χώρες όμως ε, θα ακολουθήσουν, ποια θα είναι η αλληλεγγύη των άλλων, διότι ασκείται αυτή η πίεση σε ορισμένες χώρες, στη Μάλτα και στην Ιταλία περισσότερο, όχι απαραίτητα αριθμητικά, αλλά καθαρά υπό όρους δημογραφικούς και κοινωνικούς, τι θα κάνουν οι άλλες ε, χώρες. Και και ρωτώ, άμα δεν αρχίσει να λειτουργεί αυτή η οδηγία, τι θα κάνουμε και μετά για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, ποιες είναι οι ροές που πρέπει να δεχθούμε. Τώρα εγώ αφήνω το λόγο στους άλλους ε, συναδέλφους για να μιλήσουν, αλλά εγώ είμαι πραγματικά συγκεντρωμένη στο τι συμβαίνει στην Ευρώπη, στην Μεσόγειο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συμμερίζομαι την απαγοήτευση των συναδέλφων, διότι τα συμπεράσματα δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ δεν καταλαβαίνω 7-8 χιλιάδες άτομα τα οποία έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα πρέπει να ρισκάρουν τη ζωή τους για να φτάσουν μέχρι την Ευρώπη και μετά πού θα βρούνε προστασία. Και μετά εγώ θεωρώ ότι είναι θανατηφόρο για το ευρωπαϊκό σχέδιο η Μάλτα και η Ιταλία να φορτωθούν στην πλάτη τους μονάχη τις επιπτώσεις της κατάστασης. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Δείτε τι γίνεται μεταξύ Ιταλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας. Μα πραγματικά είναι φρεχτό δηλαδή. Ε, Δοκιμάζεται το σχέδιο της ε, συμβίωσής μας στην Ευρώπη. Και πραγματικά είμαι άνω κάτω. Δεν έχουμε κανένα συμπέρασμα που να μας λέει ότι εμείς αναλαμβάνουμε εμείς παρεμβαίνουμε στη Λιβύη στρατιωτικά και μετά δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στη χώρα μας να βρούνε προστασία. Ή αυτοί που φεύγουν από την Τινησία να πούμε καθίστε εδώ δύο-τρεις μήνες, αναπνεύστε και μετά ξαναγυρίστε. Και είναι απαράδεκτο όταν μιλάμε εμείς για τη συνεργασία με την, την Ισία, για τον εκδημοκρατισμό κλπ. Να χρειάζεται να έχουμε συντονισμούς με τον κύριο Φιούλε και την κυρία Άστον. Τι θέλουν οι Τινήσοι σήμερα. Απασχόληση, μεγαλύτερους μισθούς, θα ετοιμάζουν εκλογές. Έχουμε ένα σωρό τεράστιες προκλήσεις και τι τους λέμε εμείς. Τους λέμε ορίστε ξαναπάρτε πίσω 22.000 ανθρώπους. και αυτή τη στιγμή δεν ε, ξεκινάει ο μηχανισμός ε, της ε, οδηγίας, τότε σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ότι δεν έχουμε μαζική προσέλευση. Εσείς πήγατε με το Φίλε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα η κατάσταση, ήταν πολύ πιο ε, διευρυμένη η άποψή σα και πολύ πιο λεπτή. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά ξεπερνάμε τα όρια. Εγώ πραγματικά ε, σημαίνω συναγερμό πρέπει να ξυπνήσουμε τους υπουργούς μας. Δεν μπορούμε εμεί να παίζουμε αυτό το, το, το, το άρρωστο ε, σχέδιο ανθρωπίνων ζωών μπροστά στα μάτια μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποργέτσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ εισαγωγικά να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μάλστρομ για το πώς έχει εμπλακεί σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που μας θέτει όλους, όλες τις πολιτικές δυνάμεις μπροστά σε τεράστια μηχανία πολλά από τα πολιτικά μας ε, ε, σχήματα τεινάζονται και ένας πεπισμένος ευρωσκεπτικιστής όπως είμαι εγώ που σίγουρα δεν είχε δει με καλό μάτι την οδηγία 55 στον καιρό της, σήμερα αρχίζει να αναρωτιέται για το γεγονός του πόσο δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Και τα λέω αυτά ως ευρωσκεπτικιστής. που δεν βρίσκεται λύση για το πρόβλημα. Και όλες οι Ιταλικές περιφέρειες εκτός από το αμπρούτσο λόγω των σεισμών είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους πρόσφυγες σήμερα. Αλλά άλλο πράγμα είναι οι πρόσφυγες και άλλο είναι οι δεκάδες χιλιάδες οικονομικών μεταναστών. Δείτε ποια είναι η συμπεριφορά τους. Υπάρχει μια δυσκολία των οργάνων της τάξης να τους ελέγχουν υπάρχει πρόβλημα ακόμη και στην ε, στην, ε, στον επαναπατρισμό τους ε, στην Τουνιζία. Βλέπουμε να έχουν μια πειρατική στάση τα άλλα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει ορατότητα, δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν Δηλαδή οι χώρες οι οποίες προκάλεσαν την στρατιωτική και άλλα τέτοια λένε σήμερα ότι είναι ανίκανοι να ξεκινήσουν την ε, πολιτική αλληλεγγύης και να ανοίξουν την οδηγία 55. Παρακαλώ την Επίτροπο να κάνει ό,τι μπορεί ούτως ώστε συμπαγώς και συλλογικά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση άσχετα από τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις ορισμένων ε, χωρών. Άκουσα μάλιστα την Επίτροπο να λέει η νησάκι είναι η Μάλτα. Μα αν είναι η Μάλτα νησάκι τότε η Λαμπεντούζα είναι γραμματόσημο. Είναι αδιανόητο λοιπόν να κλείσουμε εμείς μέσα σε ένα γραμματόσημο δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων με τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις που είδαμε μέχρι σήμερα. Επίσης, ε, να επικαλεστώ και την ευαισθησία αυτών που στην επιτροπή μας πάντοτε ασχολήθηκαν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. δεν ήρθε μήπως η ώρα να θεωρηθεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας όλο αυτό το εμπόριο λάθρο μεταναστών μπροστά στις τηλεοράσεις πλέον ανοιχτότατα βλέπουμε αυτούς τους ε, σωματεμπόρους τους ε, ε, οι οποίοι στα μπάρ της ακτής της Τινησίας ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους Και δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε λοιπόν αυτό το, το πράγμα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ούτως ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε και τους ε, υπεύθυνου. Ο κύριος σχετικά με την ε, επανεγκατάσταση. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ κάποια σχόλια. Ακούσαμε ότι σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε τέθη το θέμα του αν θα δέχονταν ε, κάποιου ε, παρανομού μετανάστε από την Βόρεια Αφρική που έφτασαν στην Ιταλία θα μπορούσαμε να έχουμε μια εφάνταστη αντιμετώπιση. Αντί να έρθουμε σε επαφή με τι ευρωπαϊκέ χώρε, θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή με τι βόρειο-αφρικανικέ χώρε, να του ε, ζητήσουμε να ξαναυποδεχθούν του πολίτε του. Δεν σας διάκοψα εγώ, μην με διακόπτετε και εσείς παρακαλώ. Αν υπάρχει εμφύλιος πόλεμος σε μια χώρα, θα έπρεπε να ζητήσουμε από μια γειτονική τους χώρα να τους υποδεχθεί, Μια χώρα με την οποία θα έχουν στενότερους πολιτικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικού δεσμούς, γιατί θα ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι εκεί παρά εδώ. Η κυρία Μάλιστρομ ε, είπε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε τη φήμη φρουρίου. Δεν νομίζω ότι μπορούμε όμως να κάνουμε τίποτα για να βοηθήσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε τώρα ένα πρώτο γύρο απαντήσεων στο πρώτο γύρο των ερωτήσεων και θα συνεχίσουμε μετά. Το ζήτησε και η Επίτροπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που το οργανώνετε έτσι σε γύρους ερωτήσεων για να μην χρειαστεί να απαντήσω σε 14-20 ερωτήσεις και για να μην χρειάζεται να μακρηγορήσω. Κύριε Πουσουτήλη, ναι, όντως και προς τους άλλους που το ανέφεραν υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης, αλλά τα λέτε σε λάθος θεσμικό όργανο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχώς ζητεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλληλεγγύη με την Ιταλία και μετά αλληλεγγύη με τη Μάλτα. Αλλά και αλληλεγγύη με τη Λιβύη, την Τινησία και την ε, Αίγυπτο. Περίπου 500.000 άτομα, μισό εκατομμύριο άτομα έφυγαν από τη Λιβύη. Οι περισσότεροι πήγαν στην Τινησία, κάποιοι πήγαν και στην ε, Αίγυπτο και στην ε, Τινησία και στο Τσάντ είναι μεγάλος ο αριθμός ε, των ατόμων που έχουν φτάσει στην θυσία. Πολλοί ε, ε, επέστρεψαν στις χώρες προέλευσής τους. Υπάρχουν χώρες που βοήθησαν να φτάσουν πολλοί πολίτες στις χώρες από τις οποίες προέρχονταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Καναδάς και άλλες χώρες βοήθησαν να φτάσουν στις χώρες από τις οποίες προέρχονταν πολλοί πολίτε που βρίσκονται στη Λιβύη και προέρχονται από άλλε χώρε. Υπάρχουν πρόσφυγε ε, που είναι πρόσφυγε υπό του ορισμού ε, των διεθνών οργανισμών και πρέπει να φροντίσουμε αυτού του ανθρώπου που είναι στον κατάλογο τη ε, Αρμοστία για του πρόσφυγε. Κάποιοι μπορούν να, να φτάσουν σε ορισμένε χώρε, αλλά κάποιου πρέπει να του φροντίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είπαν ότι θα δεχθούν κάποιου πρόσφυγε αλλά μιλάμε για 5.000 άτομα. Ίσως ε, λίγοι περισσότεροι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στη Λιβύη αυτή τη στιγμή, αλλά όταν μιλάμε για 5.000 άτομα ε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πρόγραμμα ε, μετεγκατάστασης και η Επιτροπή θα μπορούσε να το χρηματοδοτήσει. Σας παρακαλώ λοιπόν να συμφωνήσετε ότι είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει κανείς, αλλά μιλάμε για πράξεις κατεξουσιοδότηση και ε, συνήθως τώρα τους τελευταίους μήνες μιλάμε για την Ιταλία και ξέρουμε ότι η Λαμπεντούσα είναι ένα μικρό νησί παρότι μεταφέρονται και σε άλλα μέρη της Ιταλίας ε, οι μετανάστες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινήθηκε πολύ γρήγορα. Κάναμε την επιχείρηση εμείς που βοηθά τους συνοριοφύλακες ε, και στην Ιταλία και αλλού. Έχουμε διαθέσει κονδύλια και επίσης βοηθάμε και στην εκένωση ε, ατόμων και στη μεταφορά ατόμων από τη Λαμπεντούσα σε άλλα τμήματα της Ιταλίας. Και έχουμε πει και στην Ιταλική κυβέρνηση ότι είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε για τον επαναπατρισμό ορισμένων τυνησίων, οι οποίοι ενδεχομένως θα επιστρέψουν στην Τινησία. Ελπίζουμε ορισμένοι ε, θα αποδεχθούν κάποια προγράμματα εθελοντικού επαναπατρισμού. Οι περισσότεροι άνθρωποι από την Τινησία προέρχονται από την ίδια περιοχή που πλήττεται από ισχυρή ανεργία διότι δεν υπάρχει εισόδημα από τον τουρισμό που είχαν παλιότερα και αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιους να ξαναχτίσουν τη χώρα τους όπως είπε και ε, η κυρία Φλότχ θέλουμε να βοηθήσουμε την ανοικοδόμηση μιας νέας δημοκρατικής χώρας. Όσον αφορά το πιλωτικό πρόγραμμα για τη Μάλτα, ήταν πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραταθεί αυτό το πρόγραμμα και το κάναμε για να δείξουμε συγκεκριμένα και στην πράξη την αλληλεγγύη μα με τη Μάλτα. Μέσα σε 24 ώρε κινητοποιήσαμε περίπου 200 θέσεις, 200 άτομα που μπορούν ε, να πάνε σε άλλα κράτη-μέλη και υπάρχει και υπόσχεση για υποστήριξη από άλλα κράτη-μέλη που είπαν στην Επιτροπή ότι θα επανέλθουν και ελπίζουμε ότι θα προσφέρουν ε, κάποιες δυνατότητες για περισσότερα άτομα. Ε, Επομένω, καταλαβαίνω την έκκληση για αλληλεγγύη, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να απευθύνεται προ τα κράτη-μέλη. Για τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν, δεν προσφέρθηκαν να πάνε ούτε ένα άτομο από την Τινησία και ο μηχανισμός ε, προσωρινή προστασία είναι κάτι που μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με ειδική πλειοψηφία στα κράτη-μέλη. Μπορεί να το ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Και επίση θα πρέπει να θυμηθούμε, όπω είπε η κυρία Βίξτρομ, ότι μετά από το κοσυφοπαίδιο δημιουργήθηκε, γιατί εκατοντάδες χιλιάδων ατόμων ερχόντουσαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το ξεκινήσαμε. Και ξέρω ότι η Μάλτα είναι πολύ μικρό και ξέρω ότι και η Λαμπεντούσα είναι μικρό νησάκι, αλλά μιλάμε για 2.500 ετούντες ε, άσυλο στην Ευρώπη. Όταν μιλάμε για χίλια άτομα στη Μάλτα είναι μεγάλος ο αριθμός για τη Μάλτα, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με τα νούμερα που είχαμε σχετικά με το κοσυφοπαίδιο. Κοιτάξτε τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Εμένη, ε, Ακτή Ελεφαντοστού, Συρία. Υπάρχουν ε, πολλά ζητήματα σε πολλές γεωγραφικές περιοχές. Ας διαφυλάξουμε λοιπόν το γερό μας χαρτί για κάποια στιγμή που θα το χρειαστούμε πολύ περισσότερο. δεν έχουμε δυνατότητα να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να δεχθούν ε, άτομα, αλλά είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να υποβάλουν εκθέσεις για τη δραστηριότητά τους. Τι κάνουν δηλαδή για την υποδοχή ε, ατόμων που έρχονται από περιοχές ε, όπου υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις. Υπάρχει η Σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες που δεν μπορούν να επαναπατριστούν είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Ισχύει για ένα χρόνο και μετά επαναξιολογείται και μπορεί να δοθεί μια συνολική άδεια παραμονή για να μην περνάνε από μεμονωμένε αιτήσει ασύλου. Γίνεται μια συνολική άδεια παραμονή και πάλι χρειάζεται ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Χτες μόνο η Μάλτα και η Ιταλία το ζήτησαν, καμία άλλη χώρα. Νομίζω ότι με αυτό απάντησα σε πολλές από τις ερωτήσεις που έγιναν κονδύλια για την αλληλεγγύη. Ούτω ή άλλω, εμεί προσπαθούμε όπου μπορούμε να βρούμε κονδύλια. Στο Ταμείο Επιστροφών, στο Ταμείο για του πρόσφυγε, στο Ταμείο για τα Σύνορα υπάρχουν κάποια κονδύλια τα οποία έχουν απομείνει. Εμεί προσπαθούμε από όπου μπορούμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια. Και για αυτό που είπε ο κ. Μποργέζη για τη Λαμπεντούσα υπάρχουν στα διαθετικά ταμεία κάποια κονδύλια να βοηθήσουν τη Λαμπεντούσα να επανακτήσει την ελκυστικότητά τη για τον τουριστικό τομέα. Υπάρχουν υπάρχουν και κάποια άλλα προγράμματα στο πρόγραμμα γειτονία. Προσπαθούμε να βρούμε χρήματα όπου είναι δυνατόν, αλλά ε, όλοι γνωρίζουν περί τίνο πρόκειται. Δεν, μην νομίζετε ότι υπάρχουν εκατομμύρια κρυμμένα κάπου που ξαφνικά θα τα ανακαλύψουμε. Ξέρουμε και προσπαθούμε να τα βρούμε. Η κατάσταση είναι δύσκολη και η ύπατη αρμοστία σήμερα το πρωί ζήτησε πολλά εκατομμύρια για τον επαναπατρισμό ατόμων. Τώρα, όσον αφορά την ε, διακίνηση ε, ατόμων στην Τινησία, είναι μια πολύ υποπτή υπόθεση. Το κόστος μπορεί να είναι 1.500 ευρώ για το εισιτήριο από την Τινησία ή τις γειτονικές χώρες και είδαμε ότι τα σκάφη στα οποία μεταφέρονται είναι ιδιαίτερα επισφαλή και είναι πολύ επικίνδυνο το ταξίδι. Και βέβαια πρέπει να καταπολεμήσουμε τους διακινητές ε, ανθρώπων. Ήδη έχουν εξαρθρωθεί κάποια δίκτυα διακινητών, αλλά βεβαίω πρέπει να βοηθήσουμε προ αυτήν την κατεύθυνση και ξέρω ότι και ο Ιταλό Υπουργό ε, ζήτησε βοήθεια από αυτού. Για τον Frontex, δεν συζητήσαμε τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις για τον κανονισμό Frontex χτες. Είπαμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να έχουμε συμφωνία και με τον εισηγητή του Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να έχουμε τελικά μια συμφωνία. Και για την Eurodac δεν πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριληφθεί ε, το θέμα της πρόσβασης στην νομοθεσία, αλλά ζήτησαν και τα 27 κράτη-μέλη από την Επιτροπή να γίνει αυτό. Θα πρέπει να γίνει υπό την ευρύτερη έννοια της δέσμης μέτρων ε, και πολλοί ευρωβουλευτές, όχι όλο το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά πολλοί ευρωβουλευτές δεν συμφωνούν ιδιαίτερα, δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τον μηχανισμό του κατεπήγοντο σύμφωνα με τη σύμβαση του Δουβλίνου. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε κάποια συμβιβαστική λύση εδώ. Ελπίζω να απάντησα στι ερωτήσει σα και περιμένω και τι επόμενε ερωτήσει ε, και στι απαντήσει μου μπορεί να δώσω συμπληρωματικέ απαντήσει. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ο κατάλογο των ομιλητών ε, δεν ήταν σύντομο, αλλά διευρύνεται συνεχώ. Τώρα κλείνω τον κατάλογο των αγορητών. Σας παρακαλώ λοιπόν να μη σηκώνετε πλέον το χέρι. Έχουμε τώρα έναν δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ελπίζω να είναι και ο τελευταίος και μετά η Επίτροπος θα απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Eh, Εγώ είχα ρωτήσει τον ε, Διευθυντή κύριο Μανσερβίζη αλλά και εσείς βέβαια θα, πρέ... θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας απάντηση, οπότε θα χρειαστεί ίσως να κάνω την ίδια ερώτηση και υπό το φως βέβαια των νέων πληροφοριών που δώσατε. Καθώς εμείς μιλάμε, συνεχίζει, συνεχίζουν οι αποβάσεις. Οι μετανάστες αυτοί είτε οικονομικοί είτε πρόσφυγες άλλαξαν πλέον τις ρότες τους. Δεν πάνε στη Μάλτα πια ή στη Λαμπεντούζα, πάνε στη Λικάτα που είναι πάντα στην, εντάσσεται πάντα στην περιφέρεια του, στην επαρχία του Αγκριτζέντο. Στις 4 Απριλίου το βράδυ μετά από μία έντονη συζήτηση στην οποία και εσείς συμμετείχατε υπήρξε μία τεράστια συνένεση στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ των προσανατολισμών του Ευρωκοινοβουλίου και αυτού που αποκαλούν ορισμένοι και ίσως να μην κάνουν λάθος ε, εγωισμός των κρατών μελών δεν υπάρχουν συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, για τον επαναπατρισμό ή την επανεισδοχή. Υπάρχουν μόνο διμερείς συμφωνίες. Θα έχουμε τις επόμενες εβδομάδες ένα σχέδιο ε, αλληλεγγύης, κοινοτικής αλληλεγγύης ε, και ένα ευρωπαϊκό σχέδιο επανεισδοχής. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα είναι διαμορφωμένα όλα αυτά. Μετά από πολλές όμως συζητήσει σε μήνες, τις είχαμε. Εσείς είστε σοβαροί και τίμια ε, διανοητικά. Ε, πώς θα δώσουμε Πώς να εξοπλίσουμε εμείς όλα αυτά τα προγράμματα, με τι, με ποια χρήματα, με ποιες θετικές δράσεις. Ο Μπαρόσο πήρε και στην ε, την Ισία σήμερα. Να δούμε τι θα φέρει. Εμείς μιλήσαμε για αναθεώρηση των σχέσεων καλής γυτνίασης με τις χώρες της Μεσογείου και προβλέψαμε και περαιτέρω πόρους. Κυρία Μάλστρομ, ακούστε με τι θα γίνει. Δεν θα εφαρμόσουμε το άρθρο 55. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα αυξήσουμε τις περιπολίες, πώς θα βοηθήσουμε την Ιταλία, τη Μάλτα για τον επαναπατρισμό στη χώρα προορισμού. Σε Σίλια, αν εμείς Αν εγώ υλοποιούσα το όνειρό μου, πραγματοποιούσα το όνειρό μου να γίνω επίτροπος για τη μετανάστευση και εσείς εσύ ερχόσουν να κάνεις τον βουλευτή στη θέση μου και οι αποβάσεις αντί στην Σικελία γινόντουσαν στη Σουηδία ένα συγκεκριμένο πράγμα το οποίο θα έκανα θα ήταν να προχωρήσω με ευαισθησία όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εσύ αναφέρεις. Αλλά θα έδινα και συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, διότι αλληλεγγύη δεν υπάρχει. Η Κομισιόν έχει πίσω της μία τέρα ε, πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική εντολή, αλλά αντιμετωπίζει τους πολιτικούς εγωισμούς, τους εθνικούς εγωισμούς Πολλοί από τους συναδέλφους μου σκέφτονται τα ίδια πράγματα και ελπίζω ότι στην επόμενη συνάντησή μας θα έχουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα να πούμε. Η Επίτροπος μας ενημερώνει ότι στις 6 θα πρέπει να φύγει γιατί έχει κάποια άλλη ε, δουλειά. Είναι σαφές ότι αυτό το θέμα ε, δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε, δεν μπορούμε εδώ να καλύψουμε όλα τα σημεία, αλλά έχουμε εδώ ακόμα έναν κατάλογο ε, μελών που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις και να θέλουμε να επιτρέψουμε και στην Επίτροπο να απαντήσει. Ας πάμε λοιπόν λίγο πιο γρήγορα. Η κυρία Χιμένες Δεθερίλ, να σας ευχαριστήσω για την ε, καλή σας διάθεση. Ξεκαθαρίσαμε πολλά πράγματα, αλλά για την κατεπίγουσα κατάσταση στη Μεσόγειο, πιστεύω ότι μόνο η Κομισιόν μας δίνει πιστικές απαντήσεις. Ένα καλό πράγμα θα σας πω. Αλλά σας βλέπω πραγματικά σαν να είστε ο Δον Κιχώτης ε, που παλεύετε κατά των ανεμόμυλων. Αυτό είναι κομπλιμέντο. Ε, το πρόβλημα μεγαλώνει. Και οι βουλευτές πραγματικά έχουμε βαρεθεί να μιλάμε μόνο για την Ιταλία και μια χώρα που ήταν τόσο συσπηρωτική, ο Ντεγκάσπερ ήταν Ιταλός, να φτάνει λοιπόν αυτή η χώρα να λέει αμάν θα φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί, διότι η Ιταλική κοινή γνώμη έχει συναισθανθεί ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και εγώ επίσης όταν μιλάω με τους πολίτες ακούω αυτό το παράπονο ότι δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική και αισθάνομαι και άσχημα διότι και εγώ ως βουλευτής δεν είμαι απόλυτα πεπισμένη να τους πω ότι ναι υπάρχει αυτή η πολιτική και ο Μαρόνι με όλα όσα είπε, αυτό το οποίο είπε μόνο η κυρία Μάνστρομ σώζεται. Και σας σέβεται ιδιαίτερα διότι εκτελείται πάρα πολύ σημαντικό έργο. Αλλά όσο η Γαλλία κλείνει τα σύνορά της και θέλει μεταρρύθμιση του Σέγγεν, η Γερμανία επίσης κλείνει τα δικά της σύνορα. Θέλω να ρωτήσω την Επίτροπο, κινδυνεύει το Σέγγεν ναι ή όχι διότι τελικά την τελευταία λέξη την έχουν τα κράτη-μέλη και εμείς δεν μετράμε σε τίποτα. Θα ήθελα να ξέρω πέρα από την έλλειψη αλληλεγγύης που δίνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα προχωρήσουμε τελικά στην κοινή μεταναστευτική πολιτική. Δεν μπορούμε εμείς να ανεχόμαστε να βλέπουμε τη Μεσόγειο να μετατρέπεται σε ένα θαλασσι σε ένα θαλασσινό νεκροταφείο. Δύο λεπτά. Πολύ πιο γρήγορα θα τα πω. Διότι και εγώ συμμερίζομαι όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι για το Συμβούλιο, μα νομίζω ότι είναι σχετικά νορμάλ όλα αυτά. Διότι εμένα η αίσθηση μου είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν καμία όρεξη να βγουν από αυτό το καθεστώς της υποκρισίας το καθένας για τον εαυτό του. Ίσως θέλανε να, να λύσουν κάποια δικά τους, ε, κάποιες δικές τους διμερείς διαφορές, ίσως να κατάφεραν κάτι, αλλά δεν προχώρησαν πιο μακριά. Και αυτό γιατί σε ορισμένες χώρες υπάρχουν προεκλογικές προκλήσεις και το θέμα της μετανάστευσης δεν είναι καθόλου δημοφιλές και αφήστε δε που ενορχιστρώνεται και με τον κατάλληλο τρόπο. Δύο σύντομες ερωτήσεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα τα προσπρώξουμε εσείς και εμείς με τις καλές μας θελήσεις, πώς θα προχωρήσουμε σε μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και θα βγούμε από αυτές τις κλαδικές, τις τμηματικές πολιτικές. Πώς μπορούμε να έχουμε μια πιο πανοραμική εικόνα της μετανάστευσης. Και δεύτερο, προληπτικά Κομισιόν θα ήθελε να εκφραστεί για την αμφισβήτηση της αρχής της οικογενειακής επανένωσης και άλλων αρχών που ανέφεραν οι γαλλικές εφημερίδες, ο κύριος Σαλβάρο. Εγώ θα μιλήσω πάντως γερμανικά και όποιος θα χρειάζεται να βάλει τα ακουστικά του. Ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτής της ε, κρίσης είναι ότι τελικά σοβαρά πια αρχίζουμε να μιλάμε για μετανάστευση ότι η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί για να σεβαστεί τις, αρχι... τις αρχές της Ευρώπης. Μιλάμε για αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις. Χώρες σαν την Ιταλία Τρεις φορές τους ρώτησε η Κομισιόν. Είπε στο Μαρόνι θες βοήθεια. Όχι είπε ο Μαρόνι. Τον ξαναρώτησε θες βοήθεια. Όχι ξαναείπε. Λοιπόν και θα έπρεπε να είχε απίσει και την περηφάνεια κατά μέρο δηλαδή. Και να πει ορίστε παιδιά χρειαζόμαστε βοήθεια ήρθανε. Ήρθανε τόσοι νοματέοι, κάτι να κάνουμε, εμεί θα πάρουμε 6.000 να μοιράσουμε τους άλλους 40, δεν ξέρω τι. Αλλά αυτό δεν έγινε και το κάθε κράτος ε, μέλος ε, αρχίζει και ε, έχει μία περίεργη αίσθηση τελικά <coughs> ότι ορίστε δεν μας βοηθάνε. Ας τους δώσουμε λοιπόν αυτές τις προσωρινές άδειες παραμονής και ας πάνε όπου θέλουνε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως είπε και η συνάδελφος Φλότ, ότι αυτοί που έρχονται εδώ από την Τινησία έχουν οι άνθρωποι ανάγκη. Δεν έχουν βέβαια το δικαίωμα να τους δώσουμε πολιτικό άσυλο, αλλά έχουν ανάγκες οι άνθρωποι να τους δώσουμε τη δυνατότητα να γυρίσουν πίσω στις χώρες, στη χώρα τους. Αλλά να τους βοηθήσουμε πρώτα. Βέβαια όλοι αυτοί όταν ε, δεν είναι απαραίτητα ετούνται στο άσυλο ακόμη και όταν παίρνουν τα, τα, τους σκυλοπνίχτες για να διασχίσουν ε, την, την, την Μεσόγειο. Και τι θα κάνουμε με όλους αυτούς που παίρνουν, αναλαμβάνουν αυτόν τον κίνδυνο. Χώρες αντί Μάλτα που είναι τόσο μικρές. Και δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν σήμερα τη ρήτρα του κατεπήγοντος, αλλά δεν είναι σήμερα κατεπήγον κάτι τέτοιο. Έχετε δίκιο ότι θα ήταν περίπτωση επίγουσα ανάγκη αν ε, όλοι αυτοί ήθελαν να έρθουν ε, προ την, ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θυμάμαι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση και ξέρουμε ότι υπάρχει και πλειοψηφία στο Συμβούλιο υπέρ αυτού δεν ξέρω να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι αν είναι η Επιτροπή κατά, θα χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο για να μπορέσει να γίνει αυτή η τροποποίηση που ζητήθηκε. Σωστά? Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόκορ, δύο λεπτά. Ούτε δέκα δευτερόλεπτα δεν θέλω, Πρόεδρε. Μία ερώτηση μόνο. Βουλγαρία, Ρουμανία και Σέγγεν. Τα είπα όλα. Α, αυτή ήταν η ερώτησή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μπότσκαρτ, δύο λεπτά. Πολύ καλό το παράδειγμα του προηγούμενου ομιλητού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ συγκεκριμένη για την οδηγία σχετικά με την κακομεταχείριση των ε, παιδιών. Συζητήθηκε το θέμα ε, και της σεξουαλικής βίας ε, και θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για κακομεταχείριση παιδιών όταν διασχίσουν κάποια εθνικά σύνορα. Η έκθεση Αντζελίλη έδειξε ότι στο Κοινοβούλιο υπήρχε σαφώς πλειοψηφία υπέρ του να το συνδέσουμε αυτό το θέμα με αυτά τα οποία συμβαίνουν για αυτούς που έχουν καταδικαστεί για κακομεταχείριση παιδιών. Μιλάμε για μια προσέγγιση πρόληψης. Υπάρχει υποστήριξη από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο. Οι κάτω χώρες εξετάζουν δυνατότητες τροποποίησης και θα ήθελα να δω τι δυνατότητες υπάρχουν. Ευχαριστώ. Κύριε Σουρίτς, ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτά που μας είπατε και σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας σχετικά με την αλληλεγγύη για τους ε, ε, πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να υπάρχει κάποια ευελιξία στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και χρειαζόμαστε ε, παρεμβάσει προ τα κράτη-μέλη για να δείξουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Για το θέμα των προσφύγων, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή η Γερμανία είπε ότι μπορεί να διακόψει την ε, συμφωνία Σέγγεν και να εφαρμόσει ελέγχους στα σύνορα αν υπάρχει μια ισχυρή απειλή από την άλλη πλευρά. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει μια απειλή από την Ιταλία εφόσον η Ιταλία λέει ότι μπορεί να αρχίσει να χορηγεί θεωρήσεις διαβατηρίου ώστε να μπορούν να κινηθούν προς άλλες χώρες ε, οι ε, εισερχόμενοι από τις χώρες της ε, Βορειοαφρικής. Ε, συζητάμε τα θέματα αιτήσεων ε, ασύλου, αλλά εκτός από τους αιτούντες άσύλου έχουμε και τους οικονομικούς μετανάστες. Υπάρχουν και παραδοσιακές λύσεις μιας επιστροφής στην την Ισία, παραδείγματο χάρη. Τι άλλες λύσεις θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Διότι συνεχώς μιλάμε για έλλειψη εργατικών χεριών. Μεταξύ των προσφύγων από την Τινησία υπάρχουν πολλοί που έχουν και ακαδημαϊκά προσόντα. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για νέους πανεπιστημιακούς ούτω ώστε να δοθεί σε αυτά τα άτομα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν κάποια δυνατότητα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα αποσυμφορήσει κάπως και την αγορά στην Τινησία και ενδεχομένως θα δώσει κάποια δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά με την επανεπιστροφή αυτών των ατόμων να υπάρξουν και επαφές ε, με την ευρωπαϊκή οικονομία, να δούμε δηλαδή τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν ε, για αυτούς τους ε, οικονομικούς πρόσφυγες και όχι μόνο να προσπαθήσουμε να τους επιστρέψουμε στη χώρα προέλευσής τους. Ευχαριστώ. Κυρία Χαουμάγε. Ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστήσω ε, την ε, Επίτροπο για τις προσπάθειές της, αλλά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να πω ότι για την επανεπιστροφή θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες ε, επανεγκατάστασης ε, ε, για να δούμε αν υπάρχει κάποιο μέσο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, και να δώσουμε κάποια πρόσβαση, όπω είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, ε, σε άτομα τα οποία έχουν ε, κάποιε δυνατότητε απασχόληση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνάω τώρα στο θέμα τη Ιταλία και τη Λαμπεντούσα. Η Σουηδία είναι μικρότερη από την Ιταλία και απορροφά περισσότερου από ότι η Ιταλία. Δεν είναι ε, η μόνη χώρα, η Ιταλία, που πρέπει να απορροφήσει όλους τους πρόσφυγες στην Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία που παίρνουν περισσότερους πρόσφυγες από ότι η Ιταλία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε με ειλικρίνεια. Και το θέμα της αλληλεγγύης είναι ένα θέμα ε, ε, το οποίο μας έχει απασχολήσει και στη Γερμανία. Κάποια φορά ε, χρειάστηκε η Γερμανία να απορροφήσει 50.000 άτομα μέσα σε ένα χρόνο και δεν μας βοήθησε η Ιταλία εκείνη την εποχή. Τι μπορούμε να κάνουμε, υπάρχουν κάποιε δυνατότητε, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιε οδηγίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ισχύουν για όλε τι χώρε και χείρα βοηθείας ε, έχει δοθεί αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μαζική εισρωή προσφύγων στην Ιταλία Μπορεί να μιλάμε ε, ε, για ε, χίλια, δύο χιλιάδες και τρεις χιλιάδες άτομα στη Μάλτα που συνιστούν υπερβολικό αριθμό και θα μπορούσε να ζητήσει κανείς να βοηθήσουμε τη Μάλτα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή χώρα και έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Εκεί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αλληλεγγύη, αλλά στην περίπτωση της Ιταλίας δεν είναι το ίδιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκροτσέτα. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά και κυρίως ερωτήσεις. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Νομίζω ότι η υπεύθυνη για όλα αυτά ήταν όταν ε, αποφασίσαμε να βομβαρδίσουμε τη Λιβύη. Και λόγω αυτού του βομβαρδισμού να σας ε, να σας κάνω την ερώτηση που μου υπέβαλε ένας νέος, ένας νεαρός την Εγώ είμαι Σικελός, γνωρίζω καλά την, την μιλάω και αραβικά. Λοιπόν, λόγω αυτών των βομβαρδισμών 150 Λίβοι έφυγαν από τη Λιβύη προς την Τινησία. Με τις κινήσεις λοιπόν αυτές, ε, τις μεταναστευτικές, ήρθαν και 15.000 από αυτούς ε, στην Ιταλία. Λοιπόν έγινε η απόπειρα να κλειστεί, να κλειστεί η θάλασσα και λοιπά να μπορούν να περάσουν και τελικά η Ιταλική κυβέρνηση έδωσε, ε, έδωσε βίζες ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Εγώ ξέρετε ότι πάντοτε πίκρανα την τελική πολιτική για τη μετανάστευση. Κοιτάστε, στην Τινησία Έχουμε 800.000 με ένα εκατομμύριο κόσμο που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού. Και οι προβλέψεις από ό,τι λένε σήμερα στην Τινησία είναι χάλια για τον τουρισμό. Τι θα κάνει όλος αυτός ο κόσμος. Εμάς μας λένε τι, όταν μας λένε ορίστε πάμε να βομβαρδίσουμε όλοι τρέχουμε και βομβαρδίζουμε. Αλλά όταν πρέπει να δώσουμε ένα χέρι βάσει της πολιτικής γυτνίασης δεν το δίνουμε. Λοιπόν, πώς θα σβήσουμε εμείς τις ε, επαναστάσεις, ε, τις, επαναστα... τις αραβικές επαναστάσεις, η κυρία Αλφάνο. Λοιπόν, τη αρέσει, δεν της αρέσει, η επίτροπο, η Κακομήρα έρχεται εδώ και μας, να μας δώσει απαντήσεις ε, και την ευχαριστώ. Εγώ τώρα πιστεύω ότι το χειρότερο είναι ακόμη να έρθει διότι έχουμε χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι της ε, στη Λιβύη ε, που πήγανε από το Τσάντι ή από την Ερυθρέα και τα θύματα της, ε, του εμφυλίου θα έρθουν στην ευρωπαϊκή γη. Ρωτώ η γαλλική έλεγχη στα σύνορα είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ναι ή όχι. Και ποιοι είναι οι αντικειμενικοί όροι ούτως ώστε να αρχίσει να ισχύει η οδηγία 55. Εγώ πάντοτε άσκησα σοβαρές κριτικές στην Ιταλική πολιτική για τη μετανάστευση και ξέρω ότι η Γερμανία και η Σουηδία έχουν πολλούς μετανάστες αλλά εμείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα μέσα από το κατεπήγον πρέπει να υπάρχει μία πρόβλεψη, ένας προγραμματισμός δεν υπάρχει τελικά μεγάλη πολιτική για θέματα ασύλου ή μετανάστευσης καιρός είναι να αρχίσουμε εμείς να το λαμβάνουμε υπόψη μας και σύντομα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε εγώ ελπίζω να κάνω λάθος, άμα, αλλά άμα αρχίσουν και καταφθάνουν οι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στη Λιβύη και δεν είναι Λίβοι, τότε θα βουλιάξουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. 6 παρα 10 είναι. Κυρία Μάλστρομ, εγώ θέλω να σας συγχαρώ για όλα όσα κάνετε σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο και να σας αναφέρω το θέμα των εποχιακών αδειών παραμονής που χορηγούνται στην Ιταλία. Κοιτάξτε, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ποια είναι τα επιχειρήματα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη για να μην συμπαραταχθούν σε χώρες ε, όπως ε, η Ιταλία και η Μάλτα που αντιμετωπίζουν τις μεταναστευτικές ροές. Είπατε ότι η Γερμανία θα πάρει 100 άτομα. Οι άλλες χώρες τι θα κάνουμε, μερικέ φορές θα ήθελα να είμαι κρυμμένη κάπου στη συνεδριάση του Συμβουλίου να ακούσω την αλήθεια, να ακούω τι λένε εκεί, ο κύριο Μόλτερ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία τόμων και η Ιταλία δεν ε, ε, δίνει χορήγηση διαβατηρίου για τρεις μήνες για ανθρωπιστικούς λόγους. Τώρα κάποια κράτη-μέλη σκέφτονται να κλείσουν τα σύνορα. Σύμφωνα με την Επιτροπή είναι νομότυπα όλα αυτά. Και τέλος, πιστεύει η Επιτροπή ότι κινδυνεύει το σύστημα Σέγγεν ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Μόλντερ. Δίνω το λόγο στην Επίτροπο για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές ότι είναι δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο τώρα, αλλά και διότι δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Λιβύη και στις ε, γειτονικέ χώρες και γι' αυτό είναι δύσκολο να προετοιμαστούμε για πολλά διαφορετικά σενάρια. Όσο υπάρχει κατάσταση βία. Ε, νομίζω ότι είναι το τηλέφωνο σα Πρόεδρε. Όχι, όχι. Όσο υπάρχει βία στην ε, Λιβύη, ε, θα συνεχίσουν να φεύγουν και κάποιοι θα έρθουν και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν λοιπόν εύκολες λύσεις και αν κάποιος μα πει ότι υπάρχει κάποια εύκολη λύση, α έρθει να μας το πει να μα το τεκμηριώσει. Η Επιτροπή, όπως σα είπα, θα προτείνει στις 24 Μαου κάτι για να, κάνουμε, να υπάρξει μια συνολική λύση. Θα υποβάλουμε κάποιο έγγραφο, να δούμε ε, ε, αν μπορούμε να έχουμε κάτι σε ένα κοινό σύστημα ασύλου για τη μετανάστευση, για την καταπολέμηση τη παράνομη μετανάστευση και τη ε, διακίνηση ανθρώπων και να δούμε και δυνατότητε διευκόλυνση τη νόμιμη μετανάστευση. Τα κράτη-μέλη βεβαίω έχουν τελικά το δικαίωμα να αποφασίζουν ποιο θα μπαίνει στη χώρα τους, αλλά μπορούμε να διευκολύνουμε την νόμιμη μετανάστευση και μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλες χώρες για να το κάνουμε αυτό. Και απαντώ και στην κυρία Χίρ τώρα. Παραδείγματο χάρη μπορούμε να δούμε ποια είναι τα προσόντα των ατόμων και να βρούμε ένα πρόγραμμα που θα αντιστοιχεί στα προσόντα αυτών των ανθρώπων. Ε, υπήρχαν κάποια προγράμματα με την Τινησία στη Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά δεν έχουν λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και είναι κάτι το οποίο έχουμε αρχίσει να συζητάμε με του Τινήσου για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα. Θέλουμε να έχουμε έλεγχο των συνόρων μας, αλλά θέλουμε να βελτιώσουμε και την ένταξη των ατόμων που μπορούν νομίμως να παραμείνουν στην Ευρώπη. Μιλάμε λοιπόν για μια προσπάθεια να έχουμε μια πλήρη ολιστική εικόνα για το θέμα της μετανάστευσης. Όπως είπα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Τινησία με πολλούς τρόπους δεν έχω αριθμητικά στοιχεία για τα χρήματα, κύριε Τζακολίνη. Δεν ξέρω πόσα χρήματα έχουμε δώσει στην Τινησία. Πήγαμε για να ακούσουμε τι δικέ του προτεραιότητε, να ακούσουμε τι χρειάζονται εκείνοι. Χρειάζονται βοήθεια κατά την περίοδο των εκλογών και κατά τη δημοκρατική κατά μεταβίβαση στην δημοκρατία. Και θα πρέπει τη δική μας βοήθεια να την προσαρμόσουμε στις ανάγκες τους. Δεν έχουμε ακόμη λοιπόν αριθμητικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν κονδύλια και για την Αίγυπτο και για την Τινησία και θα δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στο ευρύτερο πλαίσιο της κινητικότητας και για θέματα ασύλου, δημιουργία πολιτικής μετανάστευσης, επιστροφών, επανεισδοχής, συνεργασία για την νόμιμη μετανάστευση και την κινητικότητα, θεωρήσεις διαβατηρίου σύντομης χρονικής διάρκειας για ορισμένες κατηγορίες ατόμων κλπ. Για την Ιταλία, όπως σας είπα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Ιταλία 171 εκατομμύρια ευρώ βρήκαμε στο Γενικό Πρόγραμμα για την Ιταλία κατά την περίοδο 2009-2011. 171 εκατομμύρια ευρώ είναι χρήματα, μεγάλο μέρος των οποίων δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την Ιταλία και βοηθάμε την Ιταλία να τα ανακατανείμει και να τα αναπροσδιορίσει για να ε, απαλύνει την ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή στη Λαμπεντούσα αλλά και σε άλλες πόλεις όπου ε, υποδέχονται μετανάστες και το συζητάμε με την Ιταλία για να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την επιστροφή των Τινησίων. Υπάρχουν και κάποιες συμφωνίες Τινησίας-Ιταλίας για τη σταδιακή επιστροφή ορισμένων ατόμων. Προς τον κύριο Μέλτε, δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει το Σέγγεν, αλλά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Υπάρχουν ελλείψεις στο σύστημα Σέγγεν το αξιολογούμε αυτή τη στιγμή. Μια επιστολή ε, υπήρχε πολύ πριν από την τωρινή ε, κατάσταση, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, υπήρχε μια επιστολή να επανεξεταστεί ο μηχανισμό Schengen. Θέλουμε να δούμε πώ μπορεί να γίνει πιο ανεξάρτητο και να βελτιωθεί ο μηχανισμό Schengen και να εξετάσουμε και τη δυνατότητα ενδεχόμενη αναστολή ε, υπό συγκεκριμένε προποθέσει. Ξέρετε ότι αν υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τη δημόσια τάξη θα μπορούσε να ανασταλεί. Θέλουμε να δούμε τώρα αν μπορεί να ανασταλεί σε περίπτωση που ένα κράτο μέλο δεν ε, σέβεται τις υποχρεώσεις του. Ε, το εξετάζουμε και ε, ξέρουμε ότι έχουν δοθεί και κάποιες προσωρινές άδειες παραμονής προσωρισμένους στην Ισίους για ανθρωπιστικούς λόγους και αυτό είναι συμβατό με το Ιταλικό δίκαιο και είναι συμβατό και με το Ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά στο Ιταλικό διάταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λέγεται ότι για να ισχύσει αυτό για όλο το χώρο Σέγγεν, αυτό είναι το άρθρο 3.2 του Ιταλικού Διατάγματος, θα πρέπει να είναι συμβατό και με την νομοθεσία σχετικά με το Σέγγεν. Δηλαδή, πρέπει κατά περίπτωση να αξιολογείται αν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα ενισχύει, αν έχουν τη δυνατότητα να επιζήσουν, αν έχουν πόρους για να επιζήσουν, αν βρίσκονται στη βάση δεδομένων CIS και υπάρχουν διάφορα κριτήρια. Αν πληρούνται όλα τα κριτήρια τότε ισχύει ε, για το Σέγγεν, διαφορετικά δεν ισχύει. Δεν έχουμε ε, δικαίωμα να κάνουμε συστηματικούς ελέγχους για το Σέγγεν, αλλά μπορούν να γίνουν μεμονωμένοι έλεγχοι με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες σε περιοχές κοντά στα σύνορα. Είναι θέμα που συζητήθηκε χθες. Ορισμένε χώρε εξέφρασαν τι ανησυχίε του επί του θέματο. Η Ιταλία προσπάθησε να καθησυχάσει τι ανησυχίε. Η Επιτροπή εξετάζει πολύ προσεκτικά την κατάσταση. Δεν μπορούμε να δράσουμε με βάση φήμε και με βάση αυτά που λένε τα μέσα ενημέρωση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποια ένδειξη παραβίαση τη ισχύουσα νομοθεσία, αλλά παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά την κατάσταση. Και προσπαθούμε να αποφύγουμε το να πολιτικοποιηθεί πάρα πολύ αυτή η συζήτηση για την πολύ σύντομη ερώτηση Σέγγεν, Βουλγαρία, Ρουμανία δεν συζητήθηκε καθόλου χτε. Αυτό είναι κάτι που είναι στα χέρια του Συμβουλίου απολύτω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Και συνεχίζονται οι συζητήσει. Ελπίζω να υπάρξει κάποια διέξοδο. Κύριε Άλβαρο, ναι. Για να αλλάξει την πρότασή της η Επιτροπή πρέπει να υπάρξει ομοφωνία. Ε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στη συνέχεια μπορούν να ε, αλλάξουν τα πράγματα, αλλά πάντως πρέπει να υπάρχει ομοφωνία. Ε, σχετικά με αυτούς που έχουν καταδικαστεί για κακομεταχείριση παιδιών είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση το θέμα, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για την επανένωση των οικογενειών. Η κυρία Γκυγιόμ έθεσε το ερώτημα. Όντως, είναι μια συζήτηση που διεξάγεται σε ορισμένα κράτη-μέλη, Γαλλία, κατοχώρες και άλλες. Υπάρχει νομοθεσία. Ο όρος οικογένεια υπάρχει σε πολλές οδηγίες και δίδεται διαφορετική ερμηνεία κάθε φορά. Καλό θα ήταν νομίζω να βρεθεί ένας κοινός ορισμός σε όλες τις οδηγίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι τώρα προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα ε, στις οδηγίες επανένωσης των οικογενειών. Αυτό δεν αφορά μόνο τους μετανάστες, αφορά ε, και ε, τα ζευγάρια ιδίου φύλου. Είναι αρκετά ευρύ λοιπόν το θέμα. Και στο τέλος του έτους θα υποβάλουμε μια πράσινη βίβλο και τώρα παρακολουθούμε τα διάφορα θέματα τα οποία θα τεθούν στην Πράσινη Βίβλο. Μπορεί να μην έχουμε εθνικά στοιχεία για πολλές χώρες, αλλά ξέρουμε ότι όντως ε, Γερμανία, Σουηδία ε, δέχονται πάρα πολλούς ε, ετούντες άσυλο αυτή τη στιγμή και σίγουρα δεν είναι η βέλτιστη κατάσταση αλληλεγγύης άμα την εξετάσουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάλμστρομ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά γιατί δεχτήκατε από 20, 20 άτομα ερωτήσεις και σχόλια εξέφρασαν τις ανησυχίες τους και ε, όπως είπατε η Επιτροπή βρίσκεται έναντι μιας δύσκολης κατάστασης και βασιζόμαστε σε εσάς να ε, σημειώσετε πρόοδο. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα περιμένουμε να ακούσουμε τα νέα σας. Σας ευχαριστούμε.